θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις από τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να μην υπάρχουν καθόλου καταχρήσεις του συστήματος. Σας ευχαριστώ κυρία Χάση. Με την παρέμβασή σας λοιπόν ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η πληροφορία, όπως είπαμε θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Συναδελφοί, η επόμενη ε, συνεδρίαση θα γίνει στις 7 Ιουλίου, αύριο δηλαδή. Ε, είναι η μέρα Σαν Φερμίν που είναι πολύ